Bien. Mes chers collègues, nous... Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ας επανέλθουμε στις εργασίες μας. Απευθύνω το καλό ορίσατε στον Επίτροπο κύριο Λεβαντόφσκι που μας κάνει την τιμή, την τιμή να συμμετάσχει στις εργασίες μας μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Προπολογισμού και τους συνεργάτες του. Στο όνομα της Επιτροπής Προπολογισμών σας εύχομαι το καλό ορίσατε και καλή χρονιά θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να συνεργαστούμε μαζί σας και για τον ετήσιο προϋπολογισμό αλλά και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιετές πλαίσιο. Θα ήθελα εκτός αυτού να απευθύνω χαιρετισμό για μικρό διάστημα στην αίθουσά μας στα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, μας τιμά ιδιαίτερος η παρουσία σας και χαιρόμαστε για αυτή την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων. Κύριε Επίτροπε, σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της επανέναρξης των εργασιών μας, ανταλλάξαμε απόψεις στα πλαίσια της Επιτροπής Ρεπολογισμών για τις δημοσιονομικές προοπτικές ευρεία ενία για τον τρόπο που εμφανίζεται ο προϋπολογισμός για το 2013. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει σε λίγες εβδομάδες αυτές τις λεγόμενες γενικές κατευθυντήρες γραμμές για τον προπολογισμό του 2013 και βεβαίως συζητήσαμε για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ή την προπαρασκευή τους για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είχατε την ευγένεια να προσκαλέσετε ε, στην προηγούμενη ε, περίοδο συνόδου του Στρασβούργου την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που διαπραγματεύεται το δημοσιονομικό πλαίσιο και στη συνέχεια αυτής της ανταλλαγής απόψεων αποφασίσαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον για μας να σας ακούσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και νομίζω ότι το απλούστερο είναι να σας παραχωρήσω το λόγο για να μας πείτε τι σας απασχολεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευγενή σας πρόσκληση και να χαιρετήσω, να ευχαριστήσω ε, και να, σε, να ευχηθώ καλές εργασίες στον προπολογισμό, καλή χρονιά. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόκλησή σας για μένα, ε, διότι δίνει την ευκαιρία να γίνουν κάποιες συζητήσεις αρχάς του ενεστώτος έτους, που θα μπορούσε να καταστεί κρίσιμη χρονιά για τα δημοσιονομικά της Ευρώπης για τον προπολογισμό. Και στο Συμβουλίο την Παρασκευή θα διεξαχθεί μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση για την προσέγγιση από κορυφή προς βάση όσον αφορά τα επίπεδα δαπανών σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά όλα την Παρασκευή. Άρα το σούτο μάλλον είναι σημαντικό να τα πούμε. Ας μην τρέχουμε αυτά την Παρασκευή. Είναι... Ε, έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη κομισιόν. την πούμε πάρα πολύ φιλόδοξα, την πούμε διπλωματικά. Οπότε ε, θα δω δύσκολα την Παρασκευή. Γι' αυτό και εγώ θα πρέπει να σας ε, πω να προβληματιστείτε σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι ρεαλιστικό για την σημερινή Ευρώπη. Για να θυμηθούμε τώρα τα βασικά μας στοιχεία. Είμεθα εξοικειωμένοι με αυτήν την προσέγγιση. Την προσέγγιση από κορυφή προς βάση. Επρόκειτο για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την σημερινή ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Είχαμε πει για το 2013 και είχαμε πει πώς θα έχουμε τη μαριθμική αναπροσαρμογή και πώς αυτό θα το προχωρήσουμε παρά τις νέες αρμοδιότητες που προσδίδει στην Ευρώπη η συνθήκη της Λισαβόνας. Και είπαμε για περισσότερο και όχι για λιγότερη Ευρώπη. Αυτό είπαμε κάνουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Να, επομένως, α, αυτός είναι ο πρώτος πυλών της προσέγγισης. Δεύτερο είναι ότι θέλουμε να έχουμε πάγωμα δύο βασικών ε, αξώνων. Ε, δαπανών, γεωργία και συνοχή. Πάμε για ένα 70% ε, μείωση ή μάλλον νέα επίπεδα και γι' αυτόν τον τρόπο ε, βλέπουμε ότι έχουμε τις νέες αυτές ε, προοπτικές, τις νέους ορίζοντες με τη δική σας ε, υποστήριξη για την διασυνοριακή εκπαιδευτική κινητικότητα, ενεργειακά δίκτυα, μεταφορά ενεργείας αλλά και τις εξωτερικές αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε για να μπορέσουμε να δώσουμε μια σωστή απάντηση στο τι πάει να πει ρεαλιστικό και τι πάει να πει φιλόδοξο θα πρέπει να δούμε ε, κάποιους, κάποιους, κάποια σημεία. Να έχουμε κάποιο μπούσουλα, κάποια σημεία αναφοράς. Αλλιώς δεν βγαίνει τίποτα όσον αφορά ε, τον ορίζοντα το που περιβάλλει αυτή, στις, ε, αυτό το όραμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές στο σημείο αναφοράς είναι η σύγκριση του ευρωπαϊκού με τους εθνικούς προπολογισμούς. Αυτό προκύπτει από κάποιο είδου φορολογική επέκταση. Νέοι περιορισμοί παρά τις διευρύνσεις. Ήδη το 2011 η επέκταση των εθνικών προπολογισμών έφτασε το 62% και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα έχουμε τα στοιχεία του 2011. Να, επομένως, πώς προκύπτει η διαφορά. Και να, πώς μπορείτε να δείτε ποιο είναι το σημείο αναφοράς. Δεύτερο δε σημείο αναφοράς είναι ε, όταν κανείς ε, αναζητεί να βρει α, ε, το τι ισχύει, θα πρέπει να κοιτάξει μια μακροπρόθεσμη τάση μέχρι το 2020 0,94% θα ενισχύσει το προπολογισμό με το GNI και σε σχέση με την επόμενη περίοδο θα είναι 1% δηλαδή μεταξύ 93 και 99 ήταν 1,18% του GNI και μεταξύ του 2000 και 2000 13 ήταν 0,62%. Δηλαδή, εν άλλες λόγες, μεταξύ του 90 και 2020 η μέση τιμή, η μέσος όγκος του προπολογισμού έπεσε κατά 20% παρά τις νέες αρμοδιότητες και παρά τις διευρύνσεις. Να, επομένως, ποια είναι τα αυθεντικά σημεία αναφοράς. Και για να ολοκληρώσουμε τον προβληματισμό μας, η απόφαση να υπάρχει σταθεροποίηση επί 7 χρόνια ε, το 2013, αυτό όφιλε να λάβει υπόψη την σημερινή συγκυρία. Τη λιτότητα και την προσπάθεια της εξυγίανση των οικονομικών σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, οι δυνατότητες ανάπτυξης δεν πρόκειται να αντικατοπτρίζονται όπως πρέπει στον ε, προπολογισμό του 2020 και σας προκαλώ να βρείτε τα άλλα παραδείγματα. Έχει ξαναγίνει αυτό σε εθνικό επίπεδο να έχουμε εκ των υστέρων εξυγίανση επί επταετία. παρά τις δέσμες μέτρων δεν πρόκειται να έχουμε την ίδια, το ίδιο φρενάρισμα στην ανάπτυξη όπως στην περίπτωση που υπάρχει αυτοσυγκράτηση σε εθνικό επίπεδο. Άρα εδώ έχουμε διαφορά και ποιοτική, όχι μόνο ποσοτική. Έχουμε μια πολυεθνική ούτω ή ε, ε, οπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο πάει παραπέρα, ξεπερνάει τα όρια αντιμετώπισης της παρούσης κρίσης. Το 2007-2013 είχαμε ε, μια αισιόδοξη Ευρώπη που αναπτυσσόταν, που πίστευε στο μέλλον της και τώρα έχουμε μια Ευρώπη της κρίσης. Να το πρόβλημα και κανείς δεν είναι από αυτό το ότι έχουμε τόσες πολλές αξιώσεις, τόσες πληρωμές σήμερα. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά όσον αφορά την μεθοδολογία για την συνεργασία, για, τις, για τις, τους προπολογισμούς. Αλλά τους τελευταίους, σε αυτές τις εβδομάδες του Δεκεμβρίου του 2011 έχουμε αξιώσεις για επιστροφές για 15 δις ευρώ. Και ενώ περιμέναμε πολύ λιγότερα. Όμως, τώρα φτάσαμε τα 15. Τις τρεις εβδομάδες του Δεκεμβρίου. Βεβαίω. Θεωρήθηκε φυσιολογικό, δεν εξέπληξε. Ε, πληρώθηκαν Τέσσερα, πέντε θα μπορούσαν να πληρωθούν εγκαίρως. αν είχαμε πόρους, πιστώσεις, αλλά δεν τις έχουμε. Άρα ξεκινούμε την νέα χρονιά με μία σόρευση μη καταβληθέντων πληρωμών. Είναι δεδομένο το έλλειμμα και το σορευμένο χρέος από το 2011 λήψη των δεουσών πληρωμών. Άρα, για να δούμε τι θα πει η, αυτή η μακρόπνοη οπτική που τώρα έχει αλλάξει. Τώρα έχουμε την συνέχιση της διαδρομής αυτής που ξεκίνησε από μια α, αισιόδοξη Ευρώπη. Όμως, τον Ιανουάριο, μετά την Πολωνική Προεδρία, έχουμε τις πραγματικές διαπραγματεύσεις για το απότερο μέλλον και δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι θα είμαστε ακόμα σε κρίση το 2020. Γι' αυτό θα ήταν αυτοκτονικό σαν ε, σενάριο για το μέλλον της Ελλάδος. Ε, επίσης και κάτι άλλο, το οποίο θα πρέπει να σας το πω με την ευκαιρία συζήτησής μας, αυτό αφορά την επενδυτική φύση του κοινοτικού προπολογισμού. Αυτό το συζητήσαμε εκτενώς, εσείς και εμείς, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι η σημερινή Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά χρειάζεται και δημόσιες επενδύσεις. Θεωρώ ότι οι επενδύσεις σε ενωσιακό επίπεδο μέσω του προπολογισμού με την συνοδεία μακροοικονομικής πειθαρχία είναι το τρομήγμα πολιτική της σημερινή Ευρώπη. Και κάποιες χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα είναι δυνατόν έτσι να επιστρέψουν στην οδό της ανάπτυξης. Να, εγωμένως, τι μπορεί να γίνει για αυτή την περίοδο μέχρι το 2020. Την συρρήκνωση στο Φρωτοτζενά έχουμε περισσότερους περιορισμού εδώ από τους εθνικούς προπολογισμούς. Τώρα έχουμε περισσότερους και έτσι έχουμε επίσης σταθερό, ένα σταθερό περιβάλλον για την Ευρώπη. περιβάλλον μέχρι το 2020. Όμως προσταθερότητα και Όλοι, όλοι συζητούν για περικοπές, είμαστε πιο στριμωγμένοι από τους εθνικούς προπολογισμούς και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από το εθνικό επίπεδο. Είναι εύκολο να λέει κανείς, κόψε, κόψε, αλλά είναι ακόμη πιο δύσκολο να συμφωνηθεί το πώς θα γίνει αυτό χωρίς να ανατρέψει την ισορροπία του προπολογισμού. Γιατί δεν προτείνουμε εμεί κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται εδώ πέρα για την καλύτερη προσφορά σε ένα παζάρι, για ένα χαλί. Πρόκειται για την μέση οδό που χαρακτηρίζεται εξόχως από ισορροπία. Και για αυτό και χρειαζόμαστε ένα αντιστάθμισμα σε αυτές τις φωνές που ζητούν περικοπές και άρα θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς την κατεύθυνση, προς την οδό της ενίσχυση της Ευρώπης και εν κατακλείδη πρέπει να σας πω ότι κατανοώ την απόψή σας για τη δική μας πρόταση. Έχουμε άλλωστε και την ε, έκθεση της Σούρα και τα πράγματα είναι δύσκολα για τους ε, ιδίους πόρους γιατί εκεί για λόγους δομής, όγκου του προπολογισμού ε, η ρύθμιση δεν είναι τόσο προφανής, όμως υπάρχει μεγάλη πίεση για το τι θα κάνει η Επιτροπή, αν θέλει, να δώσει συνέχεια στα πρόγραμμα που τρέχουν το 2013 και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να αποφύγουμε την κατάτμιση των συμφωνιών σε διαφορετικά θέματα για να μην καταστρέψουμε την ισορροπία του προϋπολογισμού και εγώ έχω διατυπώσει την ε, υπόσχεση ότι θα μείνω σταθερός στην πρόταση. Στον πρώτο γύρο επαφώνουμε το Σύμβουλο την Παρασκευή όμως χρειάζεται να ακουστεί δυνατά η φωνή μας ε, πώς δηλαδή δεν θα αποδυναμώσουμε την Ευρώπη. Πώς θα ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο το οποίο έχει φωνή όσο δυνατή χρειάζεται. Σας ευχαριστώ και πάλι την προσοχή σας και την πρόσκλησή Ευχαριστώ αγαπητέ Γιάννους. Είδατε ότι χειροκρότησε αυθόρμητα η Επιτροπή Προϋπολογισμών και επομένως δείχνει θετική ε, ε, απήχηση στα λόγια σας. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Μπέγκε. Θέλετε να μιλήσετε αμέσως Ράιμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ο Επίτροπος ήδη πριν από την πρώτη briefing συνεδρίαση με την Ιτανική Προεδρία απίθυνε ένα είδος εκκλήσεως. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι κάλεσε σε βοήθεια το Κοινοβούλιο διότι αρχίζει το έτος αυτό. Δεν έχουμε καμία αφορμή για την ώρα να αποκλίνουμε από το περιεχόμενο της διαπραγματευτικής μας εντολής ως Κοινοβούλιο που προήλθε από την έκθεση Σαλβαδόρ Γκαρίγα της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Υπάρχουν ορθοί λόγοι και μάλιστα αυτοί μόλις επαναλήφθηκαν να τηρηθεί αυτή η διαπραγματευτική μας θέση. Στους επόμενους μήνες θα εξαρτηθούν πολλά και εγώ βασίζομαι στον ρεαλισμό της Ιδανικής Προεδρίας Ας με επιτραπεί να το πω έτσι γιατί είμαι και γείτονά του. Βασίζομαι λοιπόν σε αυτό το ρεαλισμό ώστε να διεξαχθούν παράλληλες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Εάν προφανώς στο προστάδιο των διαπραγματεύσεων της Negotiation Box θα υποβληθεί στην αρχή του καλοκαιριού στο Συμβούλιο μάλλον ε, ήδη από το Μάιο θα αρχίσουν οι Υπουργοί να το συζητούν. Εγώ εκφράζω την προσδοκία πριν από αυτό να συμμετάσχουμε και εμείς στο ίδιο εντατικό διάλογο με το Συμβούλιο Υπουργών. Νομίζω ακόμη ότι θα πρέπει να λεχθεί ακόμη εν ώψη και της εμπειρίας του παρελθόντος ότι το Κοινοβούλιο έχει λάβει θέσεις και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές φλέγονται να αρχίσουν την κοινοβουλευτική του εργασία και να είναι πανέτοιμες για την διαπραγμάτευση. Διότι εάν δεν λήξουν διαπραγματεύσεις, τίποτε δεν έχει ολοκληρωθεί. Η διαπραγμάτευση δεν θα έχει λήξει. Και βέβαια η ποιότητα είναι προτιμητέα απέναντι στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο και μας ενδιαφέρει να προχωρήσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις. Αυτό όμως προϋποθέτει αυτή την παράλληλη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, διαπραγματεύσεων διότι συμφωνία, ή μάλλον διαδικασία σύμφωνης γνώμης σημαίνει απλά ότι έχουμε το δικαίωμα να πούμε ναι ή όχι στα όσα θα μας υποβάλει το Συμβούλιο. Εγώ θα προβοκάρω λίγο τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητέ Γιάννους, την προηγούμενη φορά ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου λεγόταν Γιάννους Λεβαντόσκη. Και το 2006 είχε κάνει τις σχετικές προτάσεις απέναντι στη Βρετανική Προεδρία. Τότε είχε αποτύχει ο πρώτος γύρος του Λουξεμβούργου διότι δεν είχε υπάρξει ακόμη ενία θέση στο Συμβούλιο και μετά η Κομισιόν μας πίεσε, άνωθεν μάλιστα, να δεχθούμε τα όσα εν τη σοφία του είχε εγκρίνει το Συμβούλιο και τα ποσά και τις ε, συνοδευτικές συνθήκες και όρους. Αναμένω τώρα από την σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους επιμέρους επιτρόπους από το συλλογικό όργανό τους και από τον πρόεδρο της Κομισιόν να εργαστούν στη βάση αυτής της εντολής, αυτής της εκκλήσεως και τη στιγμή που το Συμβούλιο θα πιστέψει ότι μπορεί να μας υποβάλει προσφορά χαμηλότερης ποιότητας δηλαδή κάτω από το ελάχιστον που μας εγγυάται η συνθήκη σε περίπτωση μη συμφωνίας, η Κομισιόν έρχεται να μας πει μην το δεχτείτε, απορρίψτε το, το πακέτο αυτό. Και θα ήταν καλό να λεχθεί επίσης ότι ούτε η Κομισιόν ούτε το Κοινοβούλιο θα δεχθούν οτιδήποτε είναι κάτω από τα ελάχιστα που εγγυάται η συνθήκη. Μόνο τότε και βασίζομαι ε, στην αιμονή και επιμονή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θέση αυτή. Μόνο τότε λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλφίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίασή σας και να προσθέσω δύο λόγια στα όσα είπε ο Ράιμερ μόλις και τα οποία υποστηρίζω πλήρως. Καταρχήν αναφέρατε κάποια σχόλια για την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, στο Συμβούλιο και εμείς ε, περιμένουμε με ανησυχία ε, το επόμενο πρόγραμμα του Συμβουλίου για, του Γενικών Υποθέσεων δεν ε, μπορούμε να καθορίσουμε εμεί ποια προσέγγιση θα αποφασίσουν, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να δεχτούμε επιχειρήματα που βασίζονται σε προαποφασισμένες ε, περιορισμούς. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει μαζί με τον ε, Κομισιόν να κρατήσουμε την ίδια θέση όταν θα συζητάμε τα μη δημοσιονομικά ζητήματα που θα συζητηθούν επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενους όρους που να θέσει το Συμβούλιο. Και αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ε, θα υποστήριζα πολύ και θα προωθούσα τις ε, διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές πράξεις για τις μη δημοσιονομικές προτάσεις. Μόλις κάναμε μια συνάντηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω πως αυτό θα μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εργασία μας με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε όσο γίνεται πιο δραστήριοι οι διαπραγματευτές για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τα όσα μπορούν να οριστικοποιηθούν από τις μη δημοσιονομικές προτάσεις. Έπειτα, θα υπάρξει κάποια φάση όπου θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τη διοργανική συμφωνία. Και πάλι αυτό είναι κάτι που εξαρτάται πολύ από την ε, Κομισιόν και από την πρόταση που εσείς θα υποβάλλετε. Και εφόσον υπάρχουν θέματα τα οποία συζητάμε εδώ και καιρό, θα ήθελα να προτείνω να κάνουμε κάποιες αρχικές συζητήσεις ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεων μετά με τις προτάσεις και, καταλαβα... ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι βασικές αυτές προτάσεις. Και τέλος κάτι το οποίο συζήτησα σήμερα το πρωί η Κομισιόν μπορεί να μας βοηθήσει πολύ για το θέμα των ιδίων πόρων. Καταρχήν, είναι σταθερή θέση του Κοινοβουλίου ότι αυτό δεν μπορεί να διαχωριστεί από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και η Κομισιόν θα πρέπει ρητά να το πει αυτό επίσης. Αλλά όπως ανέφερε και ο κύριος Ντεάν σήμερα το πρωί, περιμένουμε κάποιες αξιολογήσεις από πλευράς των Κομισιών και μ' άρεσε πως το από ο κύριος Ντεάν έτσι ώστε να μην υπάρξει ιδεολογική συζήτηση για τους ίδιους πόρους, αλλά να μιλήσουμε για συγκεκριμένους αριθμούς, συγκεκριμένα νούμερα. Ξέρω πως μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες στην Κομισιόν, αλλά από τη στιγμή που θα μας δώσετε υπολογισμούς επί τη βάση αυτής της πρότασης που κάνατε για τους ίδιους πόρους, τόσο καλύτερα θα είναι και για τη θέση που θα κρατήσουμε εμείς. Και επίση να μην ξεχάσουμε ότι μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να μιλήσουμε και για άλλους ίδιους πόρους, όχι σε αυτή τη φάση βεβαίως, αλλά ας δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Τελευταία μου πρόταση είναι ότι πιστεύω πως αυτή η διαδικασία και αυτό συνάδει με τα όσα είπε μόλις ο κ. Μπέγκε, ότι πρέπει να είναι δηλαδή μια ανοιχτή τελείως διαδικασία. Υπάρχει μια ομάδα ε, που, στο Συμβούλιο που λέγεται φίλοι του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και προτιμάζουν κάποιες προτάσεις που δεν είναι ανοιχτές και δεν δημοσιοποιούνται σε όλους. Εγώ θα ζητούσα από την Κομισιόν να ανοίξουμε όσο γίνεται και τις εσωτερικές συζητήσεις. Στο Κοινοβούλιο είμαστε απόλυτα διαφανείς. Να έχουμε δικούς σας εκπροσώπους εδώ, εκπροσώπους του Συμβουλίου, του, το την Προεδρία, αλλά θα θέλαμε να μπορούμε και εμείς να έχουμε πληροφορίες για τα όσα συζητώνται στο Συμβούλιο, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες μας επί τη βάση των προτάσεων που έχετε υποβάλει. Ευχαριστώ. Euh, euh, Ευχαριστώ. Οι δύο ε, για του ίδιου πόρου δεν μπορούσαν να παραβρεθούν σήμερα το απόγευμα, αλλά μα ζήτησαν να θέσουμε το εξή ερώτημα, πρόεδρε, ε, κύριε Πίτροπε. Πότε σκοπεύει η Κομισιόν να μας ε, παρουσιάσει το σχέδιο για νομικής βάσης για την δημιουργία ε, μάλλον για την χρήση ενός ποσοστού του ΦΠΑ στο προπολογισμό της Ένωσης. Γιατί έχουμε θέσει επιτάπητος δύο ε, πράγματα ως ιδίους πόρους η Κομισιόν. Ε, καταρχήν το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και δεύτερον την χορήγηση ενός τμήματος του ΦΠΑ και μας ενδιαφέρει ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα. Δίνω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους, ο Σαλβαντόρ Γκαρίγκα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι για τα όσα... Ακούσαμε και ευχαριστούμε τον κύριο Επίτροπο. Είναι πάρα πολύ σωστή η δυναμική του θέση ε, όσον αφορά τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο. Και όπως μας αναφέρει, η πιο δυναμική φωνή από θεσμικής ανήκει στο Κοινοβούλιο. Όμως, όπως ο ίδιος ε, ο εισηγητής Μπέγκε μας ανέφερε, ήδη εμείς έχουμε τοποθετηθεί στις 8 Ιουνίου πέρσι. Πρόκειται για την ε, διαπραγματευτική εντολή που έχει δοθεί ε, και πρόκειται για μια θέση που αποκρισταλώσαμε κύριε Επίτροπε η οποία πάει πολύ πιο πέρα από την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιο προχωρημένη και αυτό ακριβώς είναι κείμενο του προβλήματος ότι εμείς ε, ανέκαθεν υιοθετήσαμε μια θέση η οποία από πλευράς πολιτικής είναι ισορροπημένη όσον αφορά τις διάφορες πτέρυγες του Κοινοβουλίου, τις διαφορετικές επιτροπές, και έχουμε επομένω ε, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία οπότε και υπάρχει στήριξη, στήριξη πολιτική οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε και κάποια θέματα τεχνικά και κατα τεχνοκρατικά προτεραιότητα έχει και την παραχωρούμε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόκειται για την δομή της πρότασης και την ε, οριστική υλοποίηση του πολιετούς πλαισίου. Όμως, όσον αφορά τα βασικά αριθμητικά στοιχεία και τα ποσοστά, το θέμα ξεπερνάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δε πρόβλημα, κύριε Επίτροπε, είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής, η οποία από ό,τι φαίνεται και όπως είπατε, είναι μια πρόταση που όντως είναι ρεαλιστική και όμως το Συμβούλιο θα τη θεωρήσει μαξιμαλιστική. Θα θεωρήσω ότι μέχρι εκεί φτάνουν τα όρια. Ε, και εμείς από πλευρά μας θα είμαστε ακόμα πιο σκληροί όσον αφορά τα νούμερα και σε τέτοιο δημοτευτικό πλαίσιο θα κινηθούμε. Δεν είναι επομένως τόσο τα περιθώρια, είναι στενά. Να επομένως πώς μπορείτε να ρίξετε μια δεύτερη ματιά αναθεωρητική σε αυτή την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κατόπιν όλων αυτών ε, έχουμε το δεδομένο αυτό το πλαίσιο το οποίο θα χαρακτηρίσει τις μεταγενέστερες συζητήσεις. Και επίσης εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει να κάνετε ούτε μισό βήμα προς τα πίσω όσον αφορά τα νούμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση για νέες περικοπές. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλουμε μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση με βιώσιμο προπολισμό τα επόμενα χρόνια και κυρίω θέλουμε να ληφθούν υπόψη οι στόχοι, η στρατηγική ε, για το 2020 και εκεί πέρα θα πρέπει να κάτσουμε να σταθούμε. Επομένω, λαμβάνω υπόψη τη θέση σας, αλλά και εμείς τη δική μας, που πάει παραπέρα από τη δική σας και που εσείς ως Επίτροπος τη δική σας πρέπει και οφείλετε να την υπερσβήσετε. Γκόραν Φάρν. Thank um, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Δύο λόγια μόνο ε, σε σχέση με τόσα είπε ο Σαλβαδόρ και ο Ράινερ. Γιατί γενικά συμφωνούμε. Όμως έχω τα εξής να σας πω για τα πραγματικά περιστατικά αλλά και τα νούμερα. Θυμάστε το για το 2012 είχαμε συζητήσει πώς θα βρούμε τα σωστά στοιχεία για την εκτέλεση του προβλήματος. Επόμενος το πιο σημαντικό τώρα να κάτσουμε και να τα συζητήσουμε διότι, διότι Όπω αναφέρθηκε. Θα προσθέσει κάποια στοιχεία η Κομισιόν στο Συμβούλιο. Ε, προφανώς θα τα προσθέσουν και σε εμά. Άρα έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε την ίδια βασική πραγματεύση που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτω ώστε να μην έχουμε σύγχυση σε σχέση με το τι ισχύει και τι δεν ισχύει και να παζαρεύουμε τα ίδια. Επομένω, α δημοσιεύσουμε μερικά εξ αυτών. Όχι όλα αναγκαστικά. Να, Αυτό από εσεί στην εισήγησή σα. Διότι έτσι διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο είναι όλο συνέδριο με αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμο. Ότι ισχύει, α πούμε, α, να πάμε να βρούμε έναν Σουηδό βουλευτή και να του πούμε ότι έχει πέσει 20% ο προηγούμενο του σύστημα GNI. Θα, θα, θα, θα να με πιστέψει. Άρα θα πρέπει τα στοιχεία να δημοσιευθούν, ούτω ώστε ο κόσμο να έχει τη σωστή οπτική. Αυτό είναι το ένα που θα σα αναφέρω όσον αφορά τα νούμερα και τα πραγματικά περιστατικά. Δεύτερον τώρα, όσον αφορά το timing τα χρονικά πλαίσια γιατί γνωρίζουμε πως η Δανέζικη Προεδρία έχει τάξει κάποια χρονικά πλαίσια, περιθώρια, ε, ούτω ώστε να ξέρει πού θα κινηθεί, τι θα γίνει μέχρι τον Ιούνιο. Όμως γνωρίζουμε όλοι ότι από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του έτους αυτό είναι σαν χρόνος πάρα πολύ λίγος. Νομικές βάσεις, δύσκολα θέματα επί της αρχής, ήδη, πόρε και φυσικά τα νούμερα. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε τη σχετική ανάλυση, μια που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην υπάρχει και τόση πίεση. Ας χρησιμοποιήσουμε και την επόμενη χρονιά χρειάζεται. Πίεση θα υπάρχει από τη διοίκηση. Θα πρέπει μέχρι πρώτης πρώτου 14 να είναι όλα έτοιμα για να τα τρέξουν. Επομένως το είναι πιο σωστό, πιο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε σωστά παρά να προχωρήσουμε γρήγορα. Τελευταίο τώρα. Έχουμε τα θέματα της κάθε πολιτικής επιμέρους. Ξέρουμε το συνολικό επίπεδο των πόρων, τα θέματα της εφαρμογής. Όμως υπάρχουν και κάποια θέματα επί της αρχής. Υπάρχουν κάποια θέματα οριζόντια, αυτά που γνωρίζουμε ότι θα τα ετοιμάσει σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως την ευελιξία. Τη συζητήσαμε διαμακρών και ο Ράινερ έχει προβληματιστεί προσεκτικά για το πώς αλλιώς μπορούμε να κινηθούμε για την ευελιξία, για να μην, μείνουμε στα παραδοσιακά. Οπότε. Για κοιτάξτε, μπα και μπορούμε να φέρουμε στις τραπέζες καινούρια θέματα, ούτω ώστε να φύγουμε τι αγωνίε του παρελθόντο και να κάνουμε τι αγωνίε του Διότι το τι θα τον στον προπολογισμό, αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν για συζήτηση εδώ και δεκαετίες. Πώς θα βρεθούν περισσότεροι πόροι για ευρωπαϊκά θέματα, τα οποία είναι εκτός του προπολογισμού. Νέα χρηματοδοτικά μέσα για σημαντικά ζητήματα. Έστω και εκτός προπολογισμού. Αυτά λοιπόν να ξεκαθαριστούν τα θέματα αρχή, τα οριζόντια και όχι μόνο τα ατομιακά, κλαδικά, τα νούμερα. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Σάγκλουντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε να συζητήσετε μαζί μας αυτό το σημαντικό θέμα. Θέλω κάποια πράγματα να προσθέσω στα όσα είπαν ε, οι συνάδελφοι. Είναι καλό να βλέπει κανεί ότι το Κοινοβούλιο γενικώ ε, συμφωνεί. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που στηρίζει την διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου, πράγμα που δεν συμβαίνει στο Συμβούλιο. Αναπαρατήτως, ε, όπου βλέπουμε ότι ανάλογα με τις χώρες τα μηνύματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά και άρα οι διαπραγματεύσει ε, γίνονται πολύ πιο περίπλοκες, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις στο Συμβούλιο για τέτοια θέματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σας θυμίσω ότι παρά την καλή έκθεση ΣΟΥΡ που έγινε με καλή έκθεση ε, ε, με καλό πνεύμα συνεργαστήκαμε. Ωστόσο δεν ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε γιατί πιστεύουμε πως έπρεπε να έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα ε, κόστη, στι δαπάνες που κινούνται τις δαπάνες που στηρίζουν την ανάπτυξη. Θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε περισσότερες μεταφορές ανάμεσα στου διάφορου τομεί, πριν να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα. Μέσα περιπτώσει δεν έγινε αυτό στο βαθμό που η δική μου ομάδα θα το ήθελε. Ήθελα ωστόσο αυτό να το υπογραμμίσω γιατί στι προτάσει τη Κομισιόν το πνεύμα είναι καλό, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερα τέτοιου είδου στοιχεία γιατί η σημερινή φάση τη οικονομία θα μα αναγκάσει ούτω ή άλλω να το κάνουμε αυτό, να δούμε δηλαδή τις δαπάνες μας και να δούμε πού ακριβώς θα πρέπει να τις ε, διοχετεύσουμε. Και αυτό και με φέρνει και στα ΡΑΛ, που ίσως, ίσως ήδη γνωρίζετε, πως ε, σήμερα θα ορίσουμε έναν μόνιμο εισηγητή για τα ΡΑΛ, κάτι το οποίο επιθυμούμε στην ομάδα μας. Νομίζω πως πρέπει να γίνει μια επαρκής και ανοιχτή συζήτηση για το επίπεδο δαπάνης γιατί αυτό θα μας δείξει και πού θα μπορούσαμε να κάνουμε εξοικονομήσεις αν δεν δαπανώνται τα χρήματα και ενώ ταυτόχρονα το σύστημα είναι πολύ ευάλωτο με τα ραλ που, αναλογούν σε δύο χρόνια δαπανών. Για τους ίδιους πόρους επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας. Και είναι προφανές όταν συζητάμε αυτό το θέμα με τους εθνικούς πολιτικούς και τους υπεύθυνου για τη λήψη αποφάσεων δεν καταλαβαίνουν τι είναι ήδη οι πόροι. Δεν το καταλαβαίνουν από τεχνική άποψη και δεν καταλαβαίνουν γιατί πολλοί από εμά το βλέπουμε ως κάτι το απαραίτητο. Και πρέπει να είμαστε κάπως πιο ε, απλοί και παιδαγωγικοί σε αυτή την υπόθεση να εξηγούμε δηλαδή περί πρόκειται και η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς για τους πιθανούς ε, ίδιους πόρους γιατί έτσι οι συζητήσεις θα γίνουν πιο εύκολες και η ιδέα είναι όχι απαραίτητα να αυξηθεί το βάρος ε, το φορολογικό για τους φορολογούμενους γιατί πολλοί πολιτικοί βλέπουν ε, τους ίδιους πόρους ως νέους φόρους, ε, επιπλέον αγών φόρους και όχι όπως το βλέπουμε εμείς μέσω μιας άλλης προσέγγισης όπου τουλάχιστον ε, για τη δική μου ομάδα η προσέγγιση δεν είναι να αυξηθεί ο φόρτος της φορολογίας για τους πολίτες της Ευρώπης Ξέρω ότι με το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Θέλουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι προφανές πως θα είναι δύσκολη υπόθεση και εδώ βεβαίως αν αυτό αποτύχει, ε, η Κομισιόν θα πρέπει να μας υποστηρίξει για να αναζητήσουμε άλλες λύσεις για ίδιους πόρους, ώστε να υπάρξει αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότηση ε, του προπολογισμού της Ένωσης. Καταλαβαίνω βέβαια πως από ρεαλιστική άποψη οι ίδιοι πόροι δεν μπορούν να καλύψουν ε, όλο τον προπολογισμό, αλλά θα ελπίζω πω η Κομισιόν θα μας βοηθήσει να βρούμε μια καλή λύση. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε, η Ιζαμπέλ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα συνεχίσω με βάση τα όσα είπε ο συνάδελφος Άγγλων και άλλοι. Το ξέρουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι... Έχει ξεκινήσει από τη στρατηγική της Λισαβόνας και έχει προσθέσει τη στρατηγική 2020. Έχουμε κάνει μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και με 5% αύξηση στα ποσά του 2013 δεν θα μπορούσαμε να τα, να τα χρηματοδοτήσουμε όλα. Δηλαδή έχουμε μια μεγάλη δυσκολία και αυτό δικαιολογεί την ανάγκη ακόμη περισσότερο για ίδιου πόρου. Να προσθέσω μάλιστα ότι στο πλαίσιο αυτών των ιδίων πόρων η ιδέα είναι να γίνουν οικονομίε στου εθνικού προπολογισμού και ω προ αυτό συμφωνώ με τα όσα μα ζήτησαν οι δύο συνεισηγητέ για του ίδιου πόρου που δεν είναι παρόντε απόψε, δηλαδή την ανάγκη να έχουμε νούμερα, συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά ένα ε, ζευγάρι ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και την Κομισιόν και θέλουμε οι εθνικοί βουλευτές να μας στηρίξουν, θα έλεγα για να τους ε, ε, βάλω να τους, για να τους παροτρύνω να μας ε, στηρίξουν πόσο πολύ θα τους έδινε αυτό χώρο για τους εθνικούς ε, ε, προϋπολογισμούς γιατί θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε τα νούμερα γιατί διαφορετικά το Εθνικό Κοινοβούλια που ήδη σήμερα σε άλλα θέματα αισθάνονται παραμερισμένοι και κάποιες φορές και ξεπερασμένοι αν θέλουμε λοιπόν να τους φέρουμε κοντά μας θα πρέπει να τους δώσουμε κάποιο δόλωμα ε, αλλά και κάποια νούμερα για να τους αποδείξουμε ότι έχουν κάθε συμφέρον να παίξουν το παιχνίδι της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου από κοινού απέναντι στις δυσκολίες που θα συναντήσουμε στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ Ιζαμπέλ, ο κύριος Αρτούγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Ε, εσείς μιλήσατε για το μακροπρόθεσμο όραμα της Ένωσης. Αλλά δεν άκουσα τίποτα για όραμα. Λέτε για περικοπές. Όλο περικοπές ακούω κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο αυξάνονται οι δαπάνες. Φέτος μόνο το Συμβούλιο ανακοίνωσε περικοπές, το προσπάθησε. Όχι εσείς. Εγώ είμαι εκπρόσωπος ενός κράτους μέλους και αγωνίζομαι για τους πολίτες μου. Και πιστεύω πως ε, η ελπίδα είναι στα κράτη στα, στα κράτη-μέλη και όχι στην Κομισιόν. Δεν πιστεύω στους ίδιους πόρους, ε, με καμία δύναμη. Εθνική κυριαρχία, ναι. Είναι καιρός για αποκατάσταση στην Ευρώπη ε, και πολιτική βούληση δεν υπάρχει στην Κομισιόν. Εμείς και το κόμμα μου θα στηρίξουμε το Συμβούλιο και να αποθέτω τις ελπίδες μου σε αυτά που θα παρουσιάσει για φέτος. Merci, Monsieur Bocroche. Ευχαριστώ, κύριος Μποκρός. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή συμβολή, Γιάννος. Μια συμβολή τακτική, αν μου επιτρέπεις, για την Παρασκευή. Σε παρακαλώ μην χρησιμοποιήσεις το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊ... ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μείνει ως έχει και μάλιστα να αυξηθεί από τον πληθωρισμό γιατί δεν αυξανόταν όταν αυξήθηκαν οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Δεν είναι καλό το επιχείρημα που αντι... γιατί ε, ε, αντιλέγει το άλλο σου επιχείρημα που λέει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ διαφορετικός από τους εθνικούς. Γιατί λοιπόν να αυξάνεται ή να μειώνεται παράλληλα με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Αντί γι' αυτό έχω να σου δώσω τέσσερα άλλα, τέσσερας άλλες, ε, άλλα επιχειρήματα, άλλα, άλλη λογική. Το ένα είναι ότι ναι, καταλαβαίνουμε ότι περνάμε πολύ δύσκολο καιρό στην Ευρώπη. Ολόκληρη η Ευρώπη περνάει ύφεση και σε πολλές χώρες, είτε μας αρέσει είτε όχι, παρά τις νεοκενσιανές ε, πεπιθήσεις, οι προϋπολογισμοί δεν θα αυξηθούν. Υπάρχει ένα, ένα, μια οροφή, όχι γυάλινη οροφή, αλλά οροφή που δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, και το είπες και εσύ και πολύ το λέμε, συχνά είναι διαφορετικός στο μέγεθος και στο στόχο του. Κατά συνέπεια, ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό είναι πολύ μικρό για να συμβάλλει στην ανάπτυξη ακόμα και σε καλού καιρού. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να αυξάνεται. Και στους ε, δύσκολους καιρούς μόνο οι διορθωτικές αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη, όπως απελπισμένα προσπαθεί η Ιταλία και κάποιες άλλες χώρες. Τώρα, ως συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό, υπέρ του ευρωπαϊκού υπολογισμού, ω εξή. Ρόλο του είναι να στηρίξει αυτέ τι διαφορετικέ αλλαγέ που βοηθούν την Ευρώπη να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τη. Και ω ε, κατά συνέπεια υποστηρίζει τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει που μπορεί να επιφέρουν σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η ανεργία των νέων. Ξέρουμε ότι σε ορισμένε χώρε φτάνει ακόμα και στο 50%. Μιλάμε για τη... Μπορούμε να πούμε ότι η ανταγωνιστικότητα όχι μόνο σε επίπεδο ένωσης αλλά και παγκοσμίως αυξάνεται. Όσο εκ τούτου θα πρέπει να εντοπίσουμε κάποιες προτεραιότητες και να, το... και να προσπαθήσουμε για διευθυντικές αλλαγές εκεί, παρά να τροποποιήσουμε ολόκληρο τον ε, προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Λίγα λόγια. Πρώτα για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Είδα ένα tweet, Μάικελ, από σένα που εκφράζει την ικανοποίησή σου για τις θέσεις του Κοινοβουλίου για τις guidelines που συζητήσαμε και σήμερα το πρωί και τις τελευταίες 24 ώρες είδα και μια επιστολή που στείλατε σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα λέγοντας ότι θέλετε να μην ξεπεράσει ο προϋπολογισμός μια αύξηση του 1,9% το 2013 και να αυξηθεί το προσωπικό κατά 1% και 5% σε 5 χρόνια. Πώς θα, μάλλον να μειωθεί. Πώς θα μειωθεί το προσωπικό κατά 1% σε ένα χρόνο και 5% σε 5 χρόνια. Νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουμε με τα όσα είπατε για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο προϋπολογισμός για ανάπτυξη και δουλειές. Αυτά τα έχουμε χρησιμοποιήσει ως επιχειρήματα και στο παρελθόν τα χρησιμοποίησαμε και τα τελευταία δύο χρόνια στον γύρο του ετήσιου προϋπολογισμού και δεν μας οδήγησαν πουθενά για να επιτύχουμε δηλαδή κάτι από το Συμβούλιο. Ρωτώ λοιπόν ποια άλλα επιχειρήματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εσείς ή εμείς για να πείσουμε το Συμβούλιο και ιδιαίτερα ορισμένα στις χώρες μέλη σχετικά με τα ε, πλεονεκτήματα που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Σας ευχαριστώ. Άλλοι δεν ζητούν το λόγο. Ο λίγα σχόλια εκ μέρους μου τώρα αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Γιάννους, όπως έκαναν και οι συνάδελφοί μου, για τα νούμερα που έδωσε και τις συγκρίσεις μεταξύ των προϋπολογισμών, λαμβάνοντας υπόψη και την σύσταση βέβαια να χρησιμοποιούμε με κάποια σοφροσύνη τα νούμερα αυτά, όπως είπε και ο κ. Μπόκρος, αλλά πάντως πρόκειται για μια σύγκριση αρκετά εντυπωσιακή. Η αλήθεια είναι ότι έχοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι Τώρα, ο προϋπολογισμός της ενώσεως, αντίθετα από ό,τι λένε οι συνθήκες, χρηματοδοτείται από εθνικές συνεισφορές και αυτό σημαίνει ότι ε, πέφτει θύμα των κακών οικονομικών ε, πολιτικών ορισμένων καθαρών εισφορέων. Και εκφράσαμε την έκπληξή μας απέναντι στην αλαζονία ορισμένων χωρών που είναι αντικείμενο κακής διαχείρισης και που φορτώνουν τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κακά τους αποτελέσματα των παρελθόντων ετών. Η δυσκολία που έχουμε τα δύο όργανα μας που συνεργάζονται χέρι με χέρι είναι να επιτύχουμε ώστε το ντοσχέ αυτό όταν θα συζητηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συζητηθεί από τους ε, αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων ως αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων και όχι ως, υπουργών, ως υπουργούς οικονομικών. Και βεβαίως για να μιλάω και θα με διορθώσετε διότι στην τελευταία ε, συζήτηση είχατε ε, εσείς ηγηθεί της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου οι αρχή κατών και κυβερνήσεων στην ουσία έπαιξαν τον ρόλο λογιστών σαν Υπουργοί Οικονομικών. Είναι βέβαια ε, μικρέ οι ελπίδε μα να δούμε του υπουργού οικονομικών να άρονται στο επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Έχουμε ωστόσο την ελπίδα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να αποδειχθούν αληθινοί τέτοιοι ηγέτε πέραν δηλαδή των λογιστικών ε, συλλογισμών να λάβουν υπόψη μακροπρόθεσμα τι σημαίνει η χρηματοδότηση σε λογικό επίπεδο των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για να επανέλθει η ανταγωνιστικότητα και η χρηματοδότηση σε λογικό επίπεδο των νέων αρμοδιοτήτων που οι ίδιοι ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ε, συνθήκης Λισαβόνας που χρειάστηκε 10 χρόνια εργασιών για να καταλήξουμε σε αυτήν και τώρα δεν έχει νόημα τα επόμενα 10 χρόνια να μην δοθεί ούτε ένα ευρώ για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι αρμοδιότητες. Και εάν όπως ακόμη και αν είναι πολύ μικρός ο προϋπολογισμός όπως είπε ο Μπόκρος μπορεί μακροοικονομικά να μην μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο, μπορεί όμως να παίξει μικροοικονομικά μέσα ε, και στα πλαίσια της, αρχικής, της αρχής επικορικότητας να φροντίσει δηλαδή ώστε στην κλίμακα των 27 η αξία του δαπανόμενου χρήματος να μεγιστοποιείται με τη διαχείριση των Βρυξελών και όχι ε, σπασμένος 27 χώρες μέλη. Αυτό είναι το παιδαγωγικό επιχείρημα που πρέπει να προβάλλουμε απέναντι στους εκπροσώπους κρατών και κυβερνήσεων. Και εδώ υπάρχουν στη διαπραγμάτευση αυτή ε, τρεις μοχλοί, αν θέλετε, τρία κλειδιά. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι οι νέοι ήδη οι πόροι. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για τους νέους ίδιους πόρους, τίποτα δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Γι' αυτό και από την αρχή το Κοινοβούλιο τονίζει ότι για το ίδιο το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία επί των δαπανών, αν δεν υπάρχει συμφωνία επί των ίδιων πόρων. Το δεύτερο κλειδί είναι οι πιστώσεις πληρωμών. Εκεί το έθιξαν διάφοροι ε, συνάδελφοι, αλλά το είπατε και εσείς κύριε Επίτροπε, όταν μας αναφέρατε το τεράστιο νούμερο των πιστώσεων πληρωμών που φτάσαμε στα τέλη του, προηγούμενου, του περασμένου Δεκεμβρίου. Να γνωρίζουμε λοιπόν σαφώς ποιος είναι ο ρυθμός της κατανάλωσης, ποια είναι τα ποσά στα οποία ανέρχονται οι πιστώσεις πληρωμών μπορούν να μας πούν ότι ζητάτε διαρκώς χρήματα αλλά δεν είστε σε θέση να κάνετε τις δαπάνες. Αυτό είναι ένα απόστημα που πρέπει να σπάσει. Και ε, τρίτο, η πολιτική ικανότητα που έχουμε να θανατώσουμε αν θέλετε τις Ιερές Αγελάδες. Τουλάχιστον πάντως να τις αδυνατήσουμε. Γιατί μέσα σε ένα προπολογισμό που εν πάση περιπτώσει και παρόλες τις προσπάθειές μας δεν πρόκειται από τώρα μέχρι το 2020 να αλλάξει η τάξη μεγέθους. Έχουμε τον καθήκον μέσα στα πλαίσια αυτής της Ευρώπης που τελεί υπό κρίση να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επανέλθουμε σε ανταγωνιστικότητα. Να βάλουμε αρκετά χρήματα να φτάσουμε στην κρίσιμη μάζα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εάν κάνουμε να τα δώσουμε, να πάρουμε τα χρήματα από αλλού και να τα δώσουμε αλλού. Αυτά είναι δηλαδή τα απαραίτητα. Η πολιτική βούληση, όπως είπα, να πάρουμε από ορισμένου τομεί για να τα διαθέσουμε σε νέε πολιτικέ οι οποίε καθίσταται πολύ πιο απαραίτητε σήμερα. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα τα οποία πρέπει να θέσουμε, όπω κάναμε άλλωστε και με την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και βέβαια για τι δαπάνε που εγκρίνει η αρχή επί του προπολογισμού. Και όπω λέχθηκε ήδη, πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί της μεθόδου συνεργασίας για τις φυστώσεις πληρωμών έχουμε ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παράσχει τα στοιχεία σχετικά με το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στους διάφορους εθνικούς προϋπολογισμούς, στις χώρες μέλη δηλαδή, της υλοποίησης των νέων ιδιών πόρων, όπως είπε και η Ιζαμπέλ προηγουμένως. όσο δεν μπορούμε να δείξουμε στους εθνικούς βουλευτές αλλά και στους υπουργούς οικονομικών τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των νέων ιδίων πόρων, δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας τα πλέον αποφασιστικά επιχειρήματα. Μέσα στις συγκρίσεις, άλλωστε μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικών προϋπολογισμών, θα είναι ενδιαφέρον αν και πιο δύσκολο να γίνει, να συγκρίνουμε αυτά που πραγματικά είναι συγκρίσιμα. Είναι προφανές ότι έχουμε δαπάνες λειτουργίας πολύ μικρότερες από αυτές των εθνικών ε, κυβερνήσεων στον, εθνικό, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό η τάξη σε αυτή μεγέθου είναι περίπου 6 το 6 με 7% ενώ στι ε, ε, περιπτώσεις των εθνικών κυβερνήσεων φτάνει σε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώ διατηρούν τη δυνατότητα οι χώρε μέλη να κάνουν να έχουν και επενδυτικούς προϋπολογισμούς και πρέπει να δείξουμε στους υπουργούς οικονομικών ότι όταν προτείνουμε μία μετρίαση ορισμένων κονδυλίων δεν ερχόμαστε σε αντίφαση με αυτά που πράττουν οι ίδιοι διότι ακολουθούμε τις ίδιες γραμμές ή μάλλον αυξάνουμε τα ίδια κονδύλια που αυξάνουν και οι ίδιοι στους δικούς τους προϋπολογισμούς. Αυτά λοιπόν είναι τακτικά επιχειρήματα που βρίσκονται ότι έχουν κάποια χρησιμότητα. Θα είδατε κύριε Επίτροπε ότι η αρχική σας ομιλία προκάλεσε πολλά σχόλια και πολλές απόψεις να εκφραστούν. Uh, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ο Ράιμερ Μπέγκε είναι η ζωντανή μνήμη αυτού του σώματος του Ευρωκοινοβουλίου. αλλά οι αναμνήσεις που έχουμε από με τον Γιάν Μούλτερ και όλους όσους ε, ε, συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις από πλευράς του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικά. Αυτό που είναι διαφορά είναι ότι το κλίμα είναι πολύ πιο αρνητικό. Έχουμε πολύ περισσότερους ευρωσκεπτικιστές και περισσότερο ε, διακυβερνητική επιρροή. Θα πρέπει να είμαστε όμως πιο αισιόδοξοι για το μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Και η δεύτερη διαφορά είναι ότι από την αρχή υπάρχει κάποια μορφή συμμετοχής του Κοινοβουλίου. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα αυτής της ε, αρχικής συμμετοχής, αλλά η συνεδρία είναι την πέμπτη νομίζω για να έχουμε την πρώτη top-down συζήτηση στο Συμβούλιο. Αλλά ναι, πιθανότατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αναγκαστεί να αφήσει το ρόλο ενός ειλικρινούς ε, διαμεσολαβητή αν δούμε ότι οι αλλαγές που περνούν σε αυτή την πρόταση την, επιβα... την ε, ζημιώνουν. Όπως ξέρετε υπάρχουν κάποιες θέσεις τις οποίες θέλουμε να υπερασπιστούμε πιο έντονα και οι υπόλοιπε ε, που υπάρχουν ως ε, προσθέμενη αξία μπορεί να κοπούν από τον πρώτο γύρο. Αυτό είναι ο ρόλο τη Κομισιόν, να αγωνιστεί για μια ισορροπία στον προπολογισμό για την Ευρώπη του 2020, να μπορέσει να ανταποκριθεί στι νέε προκλήσει δηλαδή του... τη παγκόσμια κατάσταση. Και όπως ε, ακούστηκε πολλές φορές, το να κρατήσουμε ζωντανούς τους ίδιους πόρους, να ανοίξουμε το θέμα της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού είναι πολύ μεγάλη βοήθεια ε, στις διαπραγματεύσεις. Καλωσορίζουμε την στάση αυτή του Κοινοβουλίου ότι δεν επιτρέπει δηλαδή μια απλή συζήτηση για το πώς θα περικόψουμε μόνο και μόνο. Δηλαδή να υπάρχει μια συζήτηση για το μέλλον από τα δύο σκέλη του προπολογισμού. Η Δανική Προεδρία νομίζω πως το ε, Τετάρτη, την Παρασκευή, δεν θα καταλήξει συμπεράσματα, απλώς θα βολιδοσκοπήσει, θα δει ποιο είναι το κλίμα και δεν θα προβεί σε καμία τελική κρίση για το πώς θα προχωρήσουμε στα θέματα ιδίων πόρων. Θα δούμε επίσης πώς θα ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό μέσω νέων πόρων, μειώνοντας την εθνική συνεισφορά της και βοηθώντας την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών σε μια φάση λιτότητας, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό και πράγμα το οποίο αναφέρθηκε στα σχόλιά σας πολύ από τον κύριο Καλφούιν, την κυρία Ντουιρόν, τον κύριο Καλφίν ε, και όλους τους Χάγκλουντ και άλλους που μίλησαν. Ε, νομίζω όμω ότι έτσι θα μπορέσουμε να αποδώσουμε. Και για τον ΦΠΑ δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε την νομική βάση. αλλά να δούμε ποια είναι η αλλαγή του κλίματος. Εδώ και δύο χρόνια, ίσως στην πρώτη αποστολή του Αλέν Λαμασούρ, όταν έσπασε η Προεδρία, ε, όταν κόντεψε να πέσει από την καρέκλα όταν ανέφερε μία φορά τους, τους ίδιους πόρους. Βλέπουμε ότι αλλάζει το κλίμα για τους ίδιους πόρους δυναμική είναι ενδιαφέρουσα υπό την πίεση της εγχώριας πολιτικής της Γερμανίας και τους φιλελεύθερους που είναι έτοιμοι να δεχτούν ένα μικρό ε, ε, φόρο, αυτό το είδος ε, χαρτώσιμου. το κλίμα είναι λοιπόν πολύ πιο θετικό για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι ίδιοι πόροι. Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και με τον Σαλβατόρ τον Καρίγα για τη θέση του Κοινοβουλίου που είναι πολύ ξεκάθαρη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ε, τα κράτη-μέλη ώστε να μην αντικαταστήσουν την πρόταση της Κομισιόν με την άλλη πρόταση που ήταν επιτάπητος ως βάση ε, για τις διαπραγματεύσεις. και ήταν ε, κάτι παραπάνω από ό,τι οι προσδοκίες των καθαρών πληρωτών. Τώρα η Δανική Προεδρία το δέχεται αυτός μια εξορροπημένη βάση για τις διαπραγματεύσεις και επιτρέπει, προτιμά μάλλον να το συζητήσει. Αυτά. Τώρα, το δίδαγμα που αποκομίσαμε το 2012 είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν αν υπάρχει δυσπιστία για τα νούμερα τότε δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη για τις διαπραγματεύσεις. Μπορεί να χάσουμε τελείως το παιχνίδι έτσι. Είναι ευκολότερο τώρα να προχωρήσουν τα προγράμματα συνοχής αν υπάρχει λιγότερη συγχρηματοδότηση από τη δική τους πλευρά. Πρέπει να κρίνουμε ποιοι ήταν οι, πριν ήταν οι παράγοντες που επηρέασαν την απόδοση. Τα 15 δις τα Χριστούγεννα σημαίνει συγκέντρωση προβλημάτων για αυτό το έτος, το 2012. Βεβαίως ε, κατανοούμε τη θέση του Κοινοβουλίου για τον, για τον υπόλοιπο ε, προϋπολογισμό, δηλαδή οποιαδήποτε δαπάνη βρίσκεται εκτός, ε, δηλαδή αφορά τα αποθεματικά και την ευελιξία, όταν μπει στο προϋπολογισμό μπαίνει με βάση τα ίδια στάνταρ ε, εφαρμογής και ελέγχου. Αν είναι εκτός αλλά το χρησιμοποιήσουμε ως απόθεμα, ως αλληλεγγύη για τα υπόλοιπα κονδύλια άμεσα αρχίζει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες και στάνταρ εφαρμογής και ελέγχου όπως και τα άλλα είδη δαπάνης. Όμως είναι δύσκολο θέμα αυτό, το πώς θα αντιμετωπίσουμε την παραδοσιακή θέση του Κοινοβουλίου δεδομένων των περιορισμών του προϋπολογισμού. Εάν είναι μέσα, τότε μάλλον εκδιώχνει κάποια άλλα είδη δαπανών και αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα της συνοχής του προϋπολογισμού. Ξέρω ότι σε σχέση με τα όσα αναμένονταν από τον κύριο Χάγκλουντ όσον αφορά την εσωτερική μετακίνηση, αναδιάταξη προς νέες ανταγωνιστικές προκλήσεις δεν αρκεί αυτό. Ότι έπρεπε δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη, ε, με μεγαλύτερες αλλαγές από την πλευρά των εσόδων αλλά και εξελίξεις από την πλευρά των δαπανών. Ακούγοντας όμως εσάς και πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης, οι θέσεις τους είναι ε, συντηρητικές. Ακόμα και στις χώρες που κοιτούν προς το μέλλον, που είναι πιο αρωματικές, η γεωργία είναι το νούμερο ένα θέμα στα εθνικά κοινοβούλια. Και δεδομένου λοιπόν του δύσκολου, της δύσκολης εποχής δεν μπορούμε να μετακινήσουμε πολλά πράγματα. Και αυτή η θέση έχει σημασία. «207 δις στα τέλος του χρόνου, του χρόνου τα τα ραλ ε, δείχνουν ε, την απορρόφηση χρημάτων συνήθως. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις πληρωμές και τις υποχρεώσεις και παράγουμε ραλ περισσότερο όσον αφορά αυτό το κενό από όσο σε σχέση με την δυνατότητα απορρόφησης που είναι συνήθως το πρόβλημα στις αρχές των δημοσιονομικών προοπτικών ε, ίσως να μην είμαι έτοιμος να ικανοποιήσω τον κύριο Χάρτογκ με τη δική μου εικόνα για την Ευρώπη, γιατί δεν χρειάζεται να πανεφεύρουμε τον τροχό. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια στρατηγική όπου οι δαπάνες θα σχετίζονται με, την, με τα όσα έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας, στη στρατηγική 2020 δηλαδή, όσον αφορά τις περικοπές θα πρέπει να γίνονται εκεί που είναι πιο ορατές. Και ορατές είναι βέβαια οι διοικητικές δαπάνες, πτήσει τα διάφορα επιδόματα 5,6% ε, του προπολογισμού είναι οι διοικητικέ δαπάνε. Μέχρι στιγμή τα παγώνουμε όλα αυτά και ξεκινώντας το 2013 και αυτό το έχετε και στην επιστολή μου, κόβουμε και θέσεις. Κόβουμε και θέσεις, ταυτόχρονα όμως πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την Κροατία. Αυτό είναι στη συνθήκη, η Κροατία πρέπει να αντιπροσωπεύεται στο Κοινοβούλιο πρέπει να αντιπροσωπεύεται και στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους οργανισμούς. Είναι αυτό μια υποχρέωση. Θα κοστίσει 22 εκατομμύρια το 2013, ξεκινώντας τον Ιούλιο και δεν ζητάμε άλλα χρήματα παραπάνω. Έπρεπε να βρούμε εξοικονομήσεις για να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα για την Κροατία μέσα στον ίδιο προϋπολογισμό. Πολλές λοιπόν οι προσπάθειες που κάνουμε για λιτότητα ε, ο κ. Μπόκρος έσωζε την Ουγγαρία σε φάση δύσκολης οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή σου. Δεν μπορούμε πάντως να κρύψουμε τα στερεότυπα. Αν ακούσω ότι ο προπολογισμό της Ευρώπης είναι για τους ευρωκράτες, θα πρέπει να πω ότι το 94% ε, των δαπανών πάει έξω από τις Βρυξέλλες και έχει επενδυτική φύση. Και αυτό Η δυναμική του προπολογισμού μα επίσης, και αυτό είναι ένα στερεότυπο, αλλά μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει, ε, ενώ υπήρχε πολύ ανεξ, ε, ανεύθυνη δημοσιονομική πολιτική στα κράτη-μέλη. Περισσότερη Ευρώπη, αλλά λιγότερος ευρωπαϊκός, μικρότερος προϋπολογισμός ευρωπαϊκός όσον αφορά το, τη σύγκριση με το ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Αλλά βεβαίως λαμβάνω σοβαρά υπόψη τη συμβουλή σας. Το είπε και ο κύριος Μπέγκε για το πώς να ε, το περάσουμε αυτό το μήνυμα. Τι δηλαδή, ποια είναι η αξία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πέρα από τα όσα θα ακούσουμε από την Ίγκη Γκρέσλε που κατά μυστηριώδη τρόπο σιωπά ακόμα σήμερα. Η ποιότητα είναι βέβαια σημαντική. Εμείς τώρα έχουμε μπροστά μας την αλλαγή ενώ μιας κατάστασης. Δεν είναι μόνο η λιτότητα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, ναι, είναι μικρή η συμβολή, αλλά είναι σημαντική σε φάση ε, δημοσιονομικής Αν οι φτωχότερες χώρες, όπως οι βαλτικές οι χώρες, η Βουλγαρία και κάποιες άλλες, παίρνουν ε, μεταφορές κοντά στα 4-5% του ΑΕΠ. Αυτή είναι η αξία μιας ε, τέτοιας μεταφοράς. Έχει νόημα για την εθνική οικονομία και θα έλεγα ότι σε πολύ μικρότερο βαθμό μεταφορές συμβάλλουν οι αναδιατάξεις ε, συμβάλλουν στην δυναμική των χωρών αυτών. Δεν μπορούμε να το ποσοστοποιήσουμε σε κάποιο βαθμό, αλλά αυτό οφείλεται και στις, στην σωστή χρήση αυτών των κονδυλίων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα βοηθήσουν και τώρα αυτές οι συμβολές ε, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτό το πρώτο γύρο συνεργασίας για φέτος. Bien, σας ευχαριστούμε αγαπητέ Γιάννους, αγαπητέ κύριε Επίτροπε. Πραγματικά ήταν ιδιαίτερα σημαντικό που διεξαγάγαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων τώρα λίγο πριν από την επόμενη συνάντηση που θα έχουμε αύριο αντιπροσωπεία δηλαδή του Κοινοβουλίου και το τρίο των Προεδριών με παρουσία της Κομισιόν. Κοιτάζω το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε το επόμενο, έχουμε μάλλον δύο ραντεβού ε, ασυνήθι την διακοινοβουλευτική διάσκεψη που θα τελεστεί στις 27 και 28 Φεβρουαρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Επιτροπή Οικονομικών και οι Επιτροπές Οικονομικών των Εθνικών Κοινοβουλίων θα συναντηθούν για να συζητήσουν περί των δημοσιονομικών πολιτικών χωρών και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την διαπαιδαγώγηση που συζητήσαμε ήδη σήμερα. Τώρα, οι ίδιοι φορείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που εκπροσωπεί τις χώρες μέλη συναντώνται ξανά στις 22 και 23 Μαρτίου όπως είχε γίνει στις 20 Οκτωβρίου πέρσι με τη συνεργασία της Πολωνικής Προεδρίας γίνεται φέτος με τη Δανική Προεδρία όπως είπα στις 22 και 23 Μαρτίου. Αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ Γιάννους, μπορώ να σας απελευθερώσω τώρα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, τώρα θα μπορέσουμε να περάσουμε στο υπαριθμόν 15 θέμα τη ημερησία διαταξιό μα, που είναι ο κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και το καθεστώ εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής ενώσεως έχει δοθεί αυτή η έκθεση στην ε, ομάδα των φιλελευθέρων που επέλεξε ως συζητητή τον κύριο Λάιον. Κύριε Σάρφ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε, Κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή το να είναι κανείς ε, ε, μέλος αυτής της Επιτροπής και είναι μια πιο χειρές και είναι τιμή μου που με όρισε η πολιτική μου ομάδα να συνεργάζω μαζί σας και επίσης σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε ε, αντιπρόεδρο. Τώρα, για όσους δεν με γνωρίζετε, θα σας πω ότι η εμπειρογνωμοσύνη μου αφορά την Γεωργία και ε, φυσικά και γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ της ε, πολιτικής της Γεωργίας γιατί δύο χρόνια ήμουν υπουργό ή στην, ε, στην στο χαρτοφυλάκι της Γεωργίας αλλά και του προπολογισμού. Οπότε κάτι μπορώ να εισφέρω και εγώ. Οπότε τώρα αμιλητή να προχωρήσουμε στα θέματα των, των προτάσεων της Κομισιόν για τα θέματα της αλλαγής του καταστατικού που αφορά το προσωπικό και θέλω και εσείς να μου πείτε τις απόψεις σας για να δούμε μέχρι πού θέλετε να φτάσουμε. Θέλετε να φτάσουμε μόνο μέχρι το δημοσιονομική επιτυχία. Γιατί μιλάμε για ένα δις λίρες στερλίνες εξοικονόμηση μέχρι το 2020. Τα περισσότερα θα πρέπει από αυτό το 5% μίσους του προσωπικού. Επίσης, θα αλλάξει η μέθοδος υπολογισμού των επιδομάτων της ΣΑΤΑ, 65 θα πάει το όριο εξοδότησης με δυνατότητα να πηγαίνει στο 67 χωρίς μείωση των δικαιωμάτων από 37,5-40 ώρες την εβδομάδα και αλλαγές όσον αφορά τους ε, συμβασιούχους και τους όσους εργάζονται στις περιφερειακές υπηρεσίες να οι βασικές προτάσεις όσον αφορά τις προτινόμενες αλλαγές στον κανονισμό. Για να δούμε τώρα μέχρι πού θέλει να φτάσει η Επιτροπή. Στη Γιούρη το συζητήσαμε και από ό,τι έχω καταλάβει Η Επιτροπή εκείνη θα έρθει να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε εμεί τι θα κάνουμε και έχουμε τώρα και κάποια θέματα τα οποία χρήζουν διευκρινήσεω. Πρώτα-πρώτα, γιατί θεώρησε η Επιτροπή ότι οι περικοπές, οι εξοικονομήσεις θα προέλθουν από εκεί. Λάβαν υπόψη άλλα θέματα και τα απέρριψαν ου. Ας γίνει μια ανάλυση καλύτερη των σημείων από που θα προέλθουν οι οικονομίες, ιδίως όσον αφορά τις περιφερειακές υπηρεσίες. Έχει ερευνήσει η Επιτροπή το κατά πόσον ε, ε, αυτές οι αλλαγές δεν θα φύξουν κάποια προγράμματα. Επίσης, πριν το πολιετές πλαίσιο θα έχει κλείσει αυτή η συμφωνία. Ιδάλλως, τι θα κάνει η Επιτροπή. Θα αναθεωρήσει τις προτάσεις της. Θα αναζητήσει νέες λύσεις περικοπών. Τι θα γίνει με αυτούς που στεξιδοτούνται, που εκπνέουν τις συμβάσεις τους στους αντικαταστήσεις ή όχι. Και τι θα κάνει η Επιτροπή σε σχέση με τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις. Να, τι πρέπει να μας διευκρινίσει η Κομισιόν. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα, ήδη η Νομική Επιτροπή συμφώνησε ε, για το πότε θα παρουσιαστεί το σχέδιο κειμένου 1η Μαρτίου, ε, τροπολογία 8 Τρίτου, ψήφιση 26-27 Μαρτίου, άρα βουλευάς προϋπολογισμού, εμείς θα πρέπει να έχουμε την εισήγηση και συζήτηση όχι μετά τις 27 Φεβρουαρίου. 21-22 Μαρτίου να ψηφίσουμε όσον αφορά τη γνωμοδότηση και τις τροπολογίες αντιστοίχω. Άρα πάνω σε αυτά θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Μια που είναι και η πρώτη μου έκθεση εδώ, ακόμα περισσότερο έχει σημασία η γνώμη σας. Είναι και Σας ευχαριστώ. Όπως είναι γνωστό, ίσως έχω εργαστεί πολύ επί του θέματος, διότι νομίζω ότι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία με την αναδιάρθρωση αυτού του καταστατικού, όχι τόσο για να κάνουμε τις μεγάλες εξοικονομήσεις, αλλά για να διορθώσουμε ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες που δεν λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο της Κομισιόν. Δυστυχώς, δυστυχώς. Θεωρώ ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία, διότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα βαθιά ριζωμένα που θα μπορούσαν να επιληθούν. Ένα από τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα είναι ότι η αρχική μας μισθή είναι πολύ χαμηλή. Εγώ θεωρώ ότι σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα στο ελεγκτικό συνέδριο ή και στο δικαστήριο, μπορούμε να δεχθούμε να συζητήσουμε και να προσφέρουμε περισσότερα. Υπάρχουν δυνατότητες να προσφερθούν περισσότερες, καλύτερες αμοιβέ εποφελία μιας καλύτερης ε, δημόσιας υπηρεσίας. Σε άλλους τομείς θεωρώ ότι η Κομισιόν έκανε προσπάθειες. Είχα, βάλει, είχα φτιάξει ένα non-paper την προηγούμενη χρονιά, κυρίως για θέματα ελεύθερων εργασίας ημερών, ε, ταξιδιού κλπ. Και αυτά τα δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευχαριστώ. Αλλά πέραν αυτών δεν έχει γίνει τίποτα. Το 2004 ήταν η πιο πρόσφατη ε, μεταρρύθμιση του καταστατικού και εκεί προκλήθηκαν κάποιες ανισορροπίες σε βάρος των νέων χωρών μελών. Εγώ το βρίσκω αυτό κρίμα. Διότι πρέπει να επιληθούν κάποια προβλήματα και βεβαίως να εξασφαλιστεί και ίση μεταχείριση του προσωπικού και κυρίως ίση αμοιβή για ίση εργασία, διότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια άδικη μεταχείριση ανθρώπων που κάνουν την ίδια δουλειά και ωστόσο αμείβονται με 40 και 50% λιγότερα. Ένα άλλο θέμα που δεν περιλαμβάνει ε, το σχέδιο της Κομισιόν είναι κάτι που οφείλει να εξυγχρονιστεί, δηλαδή το θέμα των προαγωγών. Έχουμε κατά κανόνα προαγωγές κάθε δύο χρόνια στην επόμενη βαθμίδα. Όσο επιμελής και αν είναι κανείς, ή όσο τεμπέλης αν είναι κανείς, κάθε δύο χρόνια προάγεται αυτομάτως. Αυτό οδηγεί στην κλίμακα από ΑΔ5 μέχρι ΑΔ16 οι μόνοι που δεν προάγονται να είναι οι βουλευτές. Δηλαδή εμείς παραμένουμε για πάντα εφόρου ζωής στην ίδια βαθμίδα, όλοι οι υπόλοιποι προάγονται. Θέτω το παράδειγμα των βουλευτών επιτάπητος για να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται κάποιος εξυγχρονισμός του καθεστώτος των προαγωγών που να περιλάβει σιγά σιγά και το θέμα της επίδοσης του ε, μέλους του προσωπικού. Η συγγήτρια εδώ βαδίζει προσεκτικά. Και εγώ θα κάνω και πρόταση και για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ένα πράγμα που έκανε στην πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο σύστημα FlexiTime στην αντιστάθμιση δηλαδή του ελεύθερου χρόνου. Όποιος έχει καθήκοντα διοικητικά δεν έχει δικαίωμα στο flexi time, τα οποία ανέρχονται σε 24 μέρες συνολικά τον χρόνο, αν και δεν μπορεί να τις πάρει κανείς και τις 24 μέρες αυτές μαζί. Η Επιτροπή λέει όποιος είναι τμηματάρχης ή διευθυντής, επομένως έχει διοικητικά καθήκοντα, είτε γενικός διευθυντής είτε αναπληρωτής γενικός διευθυντής, δεν λαμβάνει πλέον αντιστάθμιση σε ελεύθερες ημέρες. Εδώ είναι ανοιχτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρόσωπα που έχουν το μισθό του διευθυντού χωρίς να έχουν τις ευθύνες του διευθυντού. Έχουμε εκεί δηλαδή το ενδεχόμενο να έχουμε έναν υπάλληλο AD9 και έναν ε, άντε 15 ο οποίο έχει ανέβει εκεί με τις προαγωγές, παίρνει τα χρήματα που παίρνει ο διευθυντή, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να συνεχίσει να παίρνει και την αντιστάθμιση σε ελεύθερε ημέρε. των υπεροριών δηλαδή. Εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι άδικο και θεωρώ ότι εδώ έχουμε το καθήκον ως μέλη της Επιτροπή Προπολογισμών να δράσουμε. Ακούστηκαν ενδιαφέροντα νούμερα σήμερα στην Νομική Επιτροπή το πρωί για την μείωση των ελεύθερων ημερών. Γιατί μια ελεύθερη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζει 20.000 ευρώ. Η μείωση αυτή θα σημάνει εξοικονομήσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ. Με όλα αυτά που συζητούνται στο επίπεδο των μισθών φτάνουμε στα 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Αλλά η μεγάλη ε, επίπτωση είναι αργότερα στις συντάξεις που φτάνει η εξοικονόμηση στα 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Εγώ νομίζω ότι αυτά πρέπει να συζητηθούν και να λυθούν και τα προβλήματα που σημειώνονται στο καταστατικό του προσωπικού. Και μιλώντας για προβλήματα θέλω να τονίσω ακόμη ότι η υπερβολική γραφειοκρατία του, καθεστώτος, του καταστατικού των βουλευτών, συγγνώμη, του, προσωπικού, του προσωπικού. Έχουμε όχι μόνο τη Γενική Διεύθυνση των ανθρώπινων πόρων, αλλά και κάθε διεύθυνση έχει τμήμα ανθρώπινων πόρων δικό της. Γιατί, εάν πάρουμε τις εκτελεστικές διατάξεις για τις άδειες και μόνο αυτές είναι 52 σελίδες. Μπορώ να σας αναφέρω στο καταστατικό, μπορώ να σας φέρω και άλλες ε, περιπτώσεις. Πραγματικά το, το, το σύστημα αποζητεί από μόνο του μια απλούστευση, μια απλοποίηση. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ούτε ξέρω πόσες ώρες περνά ο υπάλληλο ψάχνοντα το καταστατικό για να βρει πώς ρυθμίζεται η άδειά του. Έχουμε μια ευθύνη και έχουμε μια ευθύνη και απέναντι στο προσωπικό να τα φροντίσουμε αυτά και θα παρακαλέσω τον εισηγητή να δείξουμε ότι κάτι θέλουμε να κάνουμε και ότι έχουμε κατανοήσει ότι δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτε αλλά ότι είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε και τα μηνύματα που μας στέλνουν οι χώρες μέλη. Εγώ είπα μέχρι τώρα το τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σας πω τώρα κάτι για το οποίο δεν μίλησα πριν. Δεν μίλησα δηλαδή για το 16% αφορολόγητο επίδομα εκπατρισμού που λαμβάνει όλα τα μέλη του προσωπικού ακόμα και αν έχουν 20 χρόνια στις Βρυξέλλες. Και το Συμβούλιο έχει μεγάλη διάθεση να το θίξει το θέμα. Μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ επιπροσθέτως των αδειών έχει και 80, ε, και, συγγνώμη, 18, 18 ημέρες όπου είναι κλειστά τα γραφεία. Αν τα βγάλουμε αυτά, φτάνουμε σε 9 εργάσιμες ημέρες που προστίθεται στην άδεια. Όπου ένας συνήθις εργαζόμενος, αν θέλει να φύγει, για παράδειγμα μεταξύ του τέλους του έτους και της αρχής του επομένου έτους, πρέπει ο απλός εργαζόμενος να πάρει άδεια. Όμως εδώ δεν χρειάζεται. Κάθε ελεύθερη τέτοια ημέρα, κάθε τέτοια αργή εντός εισαγωγικών, ε, κοστίζει 9 εκατομμύρια ευρώ. Λέω αυτά, τα λέω αυτά γιατί πολλοί δεν τολμούν να τα θίξουν και εγώ ε, λαμβάνω πολλά εχθρικά email. Εν πάση περιπτώσει, η διεύθυνσή μου είναι γνωστή, συνεχίστε να τα στέλνετε. Χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική δημόσια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που συζητούμε τώρα δεν λύνουν το πρόβλημα. Τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε και κατεπηγόντως βάλιστα δεν έχουν γίνει. Γι' αυτό θα ήθελα να είχαμε δώσει στους εαυτούς μας περισσότερο χρόνο να εξετάσουμε δηλαδή που βρίσκονται τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν για παράδειγμα για το whistleblowing, για τις καταγγελίες. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ούτε εδώ λοιπόν υπάρχει χρόνος. Κινείται το, το, ο σιδηρόδρομος ως ταχεία και χρειάζεται να τον προλάβουμε γιατί η επόμενη φάση της τροπής του καταστατικού θα είναι πολύ αργότερα. Και ολόκληρη συζήτηση με το Συμβούλιο θα κρατήσει πολύ καιρό και θα ήταν σωστό νομίζω να ψηφίσουμε βέβαια τη γνωμοδότηση τώρα. Πάντως αρχές του καλοκαιριού να κάνουμε ένα γύρο να δούμε τι μπορεί να γίνει ως απλοποίηση του καταστατικού των υπαλλήλων. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν καλή θέληση και που ε, αναμένουν να γίνει κάτι, προτιμούν κάτι να γίνει παρά να μην γίνει τίποτα. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε ότι ο σχιώδης του ΕΛΚ θα είναι πάρα πολύ δραστήριο. Ούτω ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε σωστή προεδρία του σε αυτή την πόρτα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάρο, λέγει το λόγο. Όχι, δεν θα επανέλθω στα θέματα τη συνταγωνιστικότητα του δημοσίου. Απλώ έχω μία ερώτηση προ συζητητή και προ Επιτροπή. Ο τρόπο τη εκπροσώπηση των των υπηρεσιών, πώς θα γίνεται μια ομάδα εργασίας, ε, πώς θα γίνεται αυτό. Πώς η σχετική πρόταση έγινε δεκτή, γιατί αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε ε, και να δούμε κατά πόσον έτσι θα γίνει η προβληματική ή άλλος. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρωτώ, κύριε Γενικέ, θέλετε να λάβετε το λόγο τώρα, έχουν πολλές ερωτήσεις Δηλαδή έχετε συνεχή επαφή με εισηγητή και σκιώδης. Θέλετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, είμαστε στην διάθεση του εισηγητή. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να θυμηθούμε δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει τις προτάσεις της Επιτροπής να τις ε, εντάξουμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του καταστατικού του 2004 που ήταν πάρα πολύ ουσιαστική και που από τότε μας οδήγησε σε πάνω από δεκαετίες οικονομίες και από το 2012 θα εξοικονομούν άλλες αλλά πέντε δις μέχρι το 2020. Και φυσικά, ε, όπω είπε και η κυρία Γκρέσλε, πάρα πολύ σημαντικά είναι αυτά τα, ε, τα, θέματα. Επίση, το επίπεδο του μισθού επί την προσλήψη ε, είναι μία από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του 2004, της σχετικής αναθεώρησης. Και όσον αφορά νέους υπαλλήλου, οι οποίοι προέρχονται από κάποια κράτη-μέλη. Αυτό έχει γίνει τότε και αυτό είναι το θέμα. Επίσης άκουσα την κυρία Γκρέσλε που μας εξήγησε ότι δεν ελάβαμε υπόψη κάποια στοιχεία τα οποία εκείνη ανέφερε. Όχι, τώρα δεν είναι η ώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες. Όμως θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη κινηθεί προς ε, κάποιες κατευθύνσεις για τις προσπάθειες που ήδη έγιναν ε, το πρώτη επιτροπή μείωση προσωπικού για όλες τις ε, κατηγορίες, όχι μόνο για τους ε, διοικητικούς υπαλλήλους για κάποια κατηγορία α των υπαλλήλων πρόκειται για το σύνολο του που αμείβονται με κάποιο τρόπο, ιδίω ε, αυτοί που έχουν κάποια σύμβαση. Άρα πρόκειται για συνολική, γενική μείωση του προσωπικού που αφορά το σύνολο των θεσμικών οργάνων. Το σύνολο. Που θα οδηγήσει υποφυσιολογικές συνθήκες σε εξοικονόμηση ενός δις. Σημαντικό ποσό. Επίσης, τα είπε και ο εισηγητής ότι πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προς μια εσωτερική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών. Προς το που θα κατευθύνουν προσπάθειες, οι προσπάθειες πρόκειται να μοιραστούν μεταξύ όλων των γενικών διευθύνσεων και όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες όλες όσες έχουν διεχειριστικές αρμοδιότητες. Και αυτή η μείωση του 5% θα γίνει με ετήσιες φάσεις του 1% κάθε φορά με ε, συρρήκνωση της ιδρυτικής φάσης με μία την κατάσταση των συνταξιούχων ή τόσο πάντων την κατάσταση του ενός για κάθε δύο συνταξιούχους. 1250 πάλι λιγότερο δηλαδή την Επιτροπή. Αυτό είναι τρεις φορές το προσωπικό τη δική μου γενική διεύθυνση, κάτι το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Με αυτή την ευκαιρία επομένω. Άρα θα έχουμε τέτοιου είδου αναδιάρθρωση, τέτοιου είδου ανακατανομή του προσωπικού για αναγενική διεύθυνση και αυτό θα γίνει ανάλογα με τι προτεραιότητε που έχει τάξει η Επιτροπή. Ο επίση με αυτή την ε, ευκαιρία Πρόκειται να μειωθεί το προσωπικό εκεί όπου θεωρείται πιο λογικό. Ούτω ώστε να αναπτυχθούν, να αξιοποιηθούν οι προτεραιότητε. Τώρα, όσον αφορά την ε, δουλειά, είπαμε θα πάμε σε περισσότερε εργασίε. σε 40 ώρε εργασία. Πολλοί από του υπαλλήλου δουλεύουν περισσότερο από 40 ώρες τη βδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα... Ας μην υποτιμούμε το ότι η, αυτή η αύξηση των ορών αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Ας λάβουμε υπόψη επίσης ε, τις γυναίκες ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν, δουλεύουν 2,5 ώρες παραπάνω ε, κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τις, ε, τους παιδικούς σταθμούς κλπ. Άρα, για να επανέλθουμε σε αυτά το οποίο μας εξήγησε η κυρία Γκρέσλε, καθώς αναφορά αφορά ε, το, τις αποστολές, τα ταξίδια, εδώ η κατάσταση θα πρέπει βάθρο να αναθεωρηθεί υπό το φως των ουσιαστικών πραγματικών επιπτώσεων όσον αφορά την εξέλιξη των μέσων μεταφοράς. Από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει γίνει αναθεώρηση διότι ήταν 5-6 ώρες ο χρόνος που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο να πάει από το Παρίσι Βρυξέλλες. Τώρα χρειάζονται 2-3 ώρες. Ούτε καν αεροπλάνα δεν υπήρχαν που υπάρχουν τώρα. επομένως. θα πρέπει να κάνουμε και λάβουμε υπόψη ότι οι έξι ώρες, έξι μέρες γίνανε τρεις μέρες. Άλλαξε. Επίσης, το θέμα της ε, αποζημίωσης των σχετικών διπορικών. Και, θα βάψω αυτό που η κυρία Γκρέσλε για τις ε, προαγωγές. Θα επανέλθουμε. Τώρα όσον αφορά το flexi time. Δεν πρόκειται για μέτρο το οποίο θεσπίστηκε το 2004 στην τότε μεταρρύθμιση για να υπάρχουν περισσότερες μέρες άδεια. Και εγώ ως υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης θεωρώ ότι είναι το θέμα αυτό προφανές. Το FlexiTime θεσπίστηκε για να επιτρέψει στους υπαλλήλους ιδιαίτερα τους οικογενειάρχες να μπορούν να προσαρμόσουν την παρουσία στο χώρο εργασία ούτως ώστε να μπορέσουν καλύτερα να συνδυάσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία και τα οικογενειακά βάρη. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ συγκεκριμένε ε, κατευθύνσεις για τους ε, υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά στα τμήματα, στις διευθύνσεις κλπ. Και ρίχνοντα μια ματιά στον απολογισμό των όσων έχουν γίνει από τους διαχειριστές ανθρωπίνων πόρων, τότε δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω ότι σχετικά λίγοι υπάλληλοι χρησιμοποιούν το ρεπό που στα πλαίσια του Fixed Time δίνει την ευκαιρία κάποιος να πάρει μια μεράδια για κάποιες ε, πρόσθετε ώρε εργασία. Είναι, είναι, είναι οριακή, είναι, είναι αμιλητέ η χρήση τη δυνατότητα. Επομένω, διαπιστώθηκε ότι για τους ε, ανώτερους υπαλλήλους είπαμε δεν θα δίνεται αυτή η δυνατότητα γιατί μπορούν να διαχειριστούν τον χρόνο τους αλλιώς. για το overheads που είπε η κυρία Γκρέσλε. Κάνουμε σημαντικές προσπάθειες. Υπάρχουν εδώ πέρα ουσιαστικές ε, πρόοδοι γι' αυτό τα τις δαπάνε, δαπάνες, τα overheads. Τώρα όσον αφορά το επίδομα εκπατρισμού, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, προσλαμβάνομαι σε όλη την Ευρώπη υπαλλήλου. Και αυτό θεσπίστηκε στην αρχή γιατί δικαιολογείτο. Εμείς είπαμε ότι συνεχίζει να δικαιολογείται, αλλά θα πρέπει η συζήτηση να προχωρήσει επ' αυτού. Αυτά και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τους ανθρωπινούς πόρους, εάν θέλετε, μπορούν να απαντήσουν σε άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, σα ευχαριστώ. Και ο πρόεδρος νομίζω ότι εδώ μπορεί να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση από αυτό το σημείο. Και μήπως ο εισηγητής θέλει κάτι να πει ή να ξαγάγει ένα συμπέρασμα. Για το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τις απαντήσεις που έδωσε. Και ελπίζω να απαντηθούν και τα υπόλοιπα θα συνεχίσουμε με τους οικοδεσηγητές να δούμε και αυτοί τι θέματα έχουν τόσο να μπορέσουμε εγκαίρως να προωθήσουμε την ε, ε, έκθεση και να μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία που έταξε η νομική επιτροπή. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ και τώρα. Σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για έκθεση γνωμοδότηση όσον αφορά τις συνέπειες της δημοσιονομικές όσον αφορά την ε, αναθεώρηση του κανονισμού που διέπει το προσωπικό ε, είμαστε συναρμόδιοι εμεί και η Νομική Επιτροπή. Και σα πενθυμίζω το, το, το, το, χρονοδιάγραμμα που στο COP News δεν αναφέρεται, αλλά λέει, ε, αφορά την, ε, τον εισηγητή. 8, Φεβρουαρίου θα έχουμε το κείμενο για μετάφραση. Στην Νομική Επιτροπή θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση τροπολογιών 26-27 Μαρτίου και η ψήφιση θα γίνει τον Απρίλιο. Τώρα, όσον αφορά τη δική μας ε, γνωμοδότηση, θα ψηφίσουμε 21-22 Μαρτίου. Δηλαδή, μία εβδομάδα πριν την Νομική Επιτροπή. Και και ο Φεβρουαρίου πρόκειται να οριστικά ή το κείμενο του συνάδελφου Λάιμ. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Και τώρα, το τελευταίο θέμα είναι το 16. Αφορά την εταιρική σχέση, την συμφωνία, την αλληλευτική με την Μοζαμβίκη. Πρόκειται για μια αλληλευτική συμφωνία τριετή με την Δημοκρατία του Ισμοζαμβίκης. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό. Μικρή αλληλευτική συμφωνία που δεν δεσμεύει και πολύ. Τα οικονομικά του της Ένωσης. Να πω ότι τον Ιανουάριο του 2012 ξεκινάμε και εξετάζουμε μια ε, έκθεση για μια συμφωνία που αρχίζει να ισχύει από την 1η, 1η 12. Ε, δηλαδή πρέπει πρώτα να τη συζητήσουμε ενώ ήδη πρέπει, έπρεπε να έχει αρχίσει να ισχύει. Ε, βέβαια υπάρχουν και χειρότερα. Υπήρχαν και συμφωνίες που τις διαπραγματευτήκαμε αφού είχαν ήδη αλλιευθεί τα ψάρια. Μπας περιπτώσει. Πρέπει κάνουμε, να κάνουμε αυτή τη διαπίστωση. Τώρα, για την Μοζαμβίκη και το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας υπάρχουν πολλές σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με προηγούμενες συμφωνίε που μας είχαν υποβληθεί ε, και μάλιστα διπλασιάζεται σχεδόν ε, το ποσό που αφιερώνεται στην ανάπτυξη της παλευτικής της τοπικής αλληλευτικής πολιτικής έτσι ώστε να μπορούν ε, οι Μοζαμβικανοί να ψαρεύουν τα ψάρια που κυκλοφορούν στη δική τους, ε, στα δικά τους αλληλευτικά ε, ύδατα. Επιπλέον προστατεύονται οι αλληλευτικοί πόροι, υπάρχουν εκεί οικολογικά προγράμματα αλλά και πειρατεία. Και όπως φαντάζεστε η ομάδα μας χαίρεται για την προστασία των αλληλευτικών πόρων. Αν και λοιπόν σε αυτές τις ελευτικές συμφωνίες υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα, ότι δηλαδή μπορεί να αναθεωρηθούν προς τα πάνω αν το επιτρέπουν οι συνθήκες ε, όσον αφορά τους όρους και τη συμφωνία. Εδώ δεδομένες της μικρής κλίμακας συμφωνίας οι αλλαγές δεν πρόκειται να είναι τέτοιες που να μας ενοχλήσουν για να συνεχίσουμε μια ενδεχόμενη αύξηση. Ε, για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν είμαστε υπέρ αυτής της συμφωνίας και επιθυμούμε να εθαρρύνουμε την Κομισιόν για να κάνει τέτοιου είδους συμφωνίες που στο μέλλον θα είναι πιο έγκαιρα, θα υποβάλλονται πιο έγκαιρα και ακόμα θα είναι και το περιεχόμενο τους καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γκρελιέ. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος Αλφονσί. Ε, θα ήθελα μόνο δύο διευκρινήσεις. Το ποσό της οικονομικής αντιστάθμισης της ετήσιας ε, φαίνεται να είναι χαμηλότερο από ό,τι παλιότερα, αλλά είναι πολύ ψηλό σε σχέση με τον όγκο των αλλιευμάτων σε αυτό το τομέα. Έπειτα, το ποσό που δίνεται για την αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό περνά από τις 270, ε, από τις 270 στις 460.000 ευρώ. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Très bien, je vous remercie. Σας ευχαριστώ και εάν δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο, να θυμίσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 16 Η Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού είναι στι αρχέ του Μαρτίου, ώστε η Επιτροπή Αλληλεία να ψηφίσει το Μάρτιο, μέσα στο Μάρτιο και στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε με τέσσερι μήνε καθυστέρηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο λιγότερο άσχημα από ό,τι προηγούμενα έτη, αν κατάλαβα καλά τα όσα είπε με χιούμορ, ο εισηγητή. Μπορεί να απαντήσει η Κομισιόν στην ερώτηση που τη έθεσε. Αν μπορεί τώρα, α το κάνει αργότερα. Αλλά, εν περιπτώσει, για να μην έχουμε την εντύπωση ότι μόνοι μας προσπαθούμε. Θα έχετε γραπτή απάντηση από την Κομισιόν, μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Εξαντλήσαμε την ημερήσια μας διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν διάφορα, ε, λίγες συνεδρίες, αλλά θα κρατήσω για λίγα λεπτά στην αίθουσα τους συντονιστές. Θα έχουμε μια σύντομη συνεδρίαση των συντονιστών και ζητώ και από τους διερμηνείς να μείνουν μαζί μας κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, ώστε να μας διευκολύνουν. Διακοπή 5 λεπτών.